ενημέρωσε λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το άρθρο, η διάσκεψη των Προέδρων ότι έχουμε κάποιες... Ε, έχουμε ένα αίτημα της Επιτροπής ΕΚΟΝ, στο οποίο δεν υπήρχε κάποια αντίρρηση από την διάσκεψη των Προέδρων. Εάν δεν υπάρχει κάποια πολιτική ομάδα ή 40 ευρωβουλευτές οι οποίοι θα απορρίψουν το αίτημα αυτό, τότε το αίτημα εγκρίνεται. Αλλιώς θα πρέπει να ψηφίσουμε. Υπάρχει βεβαίως το σχέδιο στο site του Κοινοβουλίου. Τώρα περνάμε στη δήλωση της Κομισιόν για την απόφαση